και να μην μείνει απομακρυσμένη από τους πολίτες της. Ευχαριστώ. Uh, uh, thank you. Thank you. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση, η σύντομη αυτή συζήτηση για τις ε, πλημμύρες στην Ευρώπη φέτος. Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej. Και τώρα, όπω προβλέπει η μερίσια διάταξη, θα έχουμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δεκάτη επέτειο του ψηφίσματος ε, των ε, Ηνωμένων Εθνών, το υπαριθμό 1325, για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Καλωσορίζω τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα δώσω πρώτα το λόγο στον ε, κύριο Ολιβιέ Σαστέλ από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι βουλευτές. Έχω την τιμή να λαμβάνω το λόγο σε μία συζήτηση εκπροσωπώντας την είπατε εκπρόσωπο τη Λελδιάστον. Επιτρέψατε μου καταρχάς ε, κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ενδιαφέρον, το μόνιμο ενδιαφέρον που επιδεικνύει για ε, τις γυναίκες, την υγεία και τη, την ειρήνη και την ασφάλεια. Και να υπενθυμίσω όπως γνωρίζετε άλλωστε και εσείς ότι το Κοινοβούλιο ήταν το πρώτο ε, θεσμικό όργανο ένα μήνα μόνο μετά την έγκριση του ψηφίσματος 1325 που ζήτησε την υιοθέτησή του μέσω ψηφίσματος ψηφίσματο του Κοινοβουλίου βέβαια. Δέκα χρόνια μετά μπορούμε μόνο πρόοδου να διαπιστώσουμε. Ήδη υπάρχει ένα διεθνέ ε, πλαίσιο το οποίο έχει ενισχυθεί σημαντικά ιδίω μετά την ε, έγκριση το 2009 ε, των ψηφισμάτων 1888 και 1889. Έχουμε και ε, εκπρόσωπο ειδικό ε, για τη θέση των γυναικών σε ένοπλε συγκρούσει ε, και αυτό αποτέλεσε επίση ένα σημαντικό βήμα. Επίση υπάρχουν σήμερα πάνω από 20 εθνικά σχέδια ανά τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, παρ όλα αυτά η κατάσταση εξακολουθεί να υπάρχει αυτή. Και γι' αυτό η πραγματικότητα υπαγορεύει την ανάγκη προστασίας των γυναικών, την συμπερίληψη τη διάστασης αυτής για τι ειρηνευτικέ διαδικασίες που μέχρι στιγμή ε, υπολείπεται. Έχουμε βία κατά των γυναικών, κατά των νεαρών κοριτσιών, ιδίω σεξουαλική και σεξουαλική κακοποίηση που στοιχίζει και ζωές ε, βέβαια και αυτό σε πλήρες ε, καθεστώς ατιμορρησίας σε πολλές περιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, αμετακίνητα δεσμευμένη στην εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 και των επακόλουθων ψηφισμάτων. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας μία στέρη, με εύρωστη πολιτική για τις γυναίκες στην ειρήνη και την ασφάλεια που καλύπτει όλες τις σχέσεις των εξωτερικών, όλες τις πτυχές των εξωτερικών σχέσεων μεταξύ αυτών και την αναπτυξιακή συνεργασία. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω κάποια συγκεκριμένα επιτεύγματα. Μία από τις ε, δράσεις είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών. Προς το στόχο αυτό, οι εμπειρογνώμονες των θεσμικών οργάνων των κρατών μελών ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν σε μια ειδική ομάδα, Task Force. Έχουν αυξηθεί τα προγράμματα σε εθνικό επίπεδο. Δέκα κράτη-μέλη έχουν εθνικό σχέδιο δράσης αυτή τη στιγμή και άλλα δύο είναι σε εξέλιξη, σε προετοιμασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στη διάθεσή της επίσης κάποια προγράμματα τα οποία τα αποκρίνονται στις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών ε, σε καταστάσεις ενόπλων συγκρούσεων αλλά και μετά την επίλυσή τους. Παροχή ιατρικών υπηρεσιών επίσης σε θύματα σεξουαλικής βίας. Μέσα σε δύο χρόνια χρηματοδοτήθηκαν ε, προγράμματα σε 67 χρόνια. Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ ήταν ο προπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να χρησιμοποιεί ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση των πτυχών του φύλου ε, σε αυτά τα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας. Η Ένωση διαθέτει κάποια σημεία επαφή, συμβούλους για ζητήματα φύλου στις 13 ε, πολιτικής, ε, της κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και οι δύο σημεία επαφή σε θέματα φύλου σε πάνω από 80 αντιπροσωπείες παγκοσμίω. Και αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή κάνουμε είναι να ολοκληρώσουμε την έκθεση η οποία μιλά για τις πτυχές του φύλου και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πώς αυτά εντάσσονται στην πολιτική, ε, στην ΚΕΠΑ. Επίσης συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στενά με την κοινωνία των πολιτών για να ευνοήσει τη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας. Για το 2011 προβλέπουμε ειδικά σχέδια για την υποστήριξη δικτύων γυναικών σε χώρες που πλήττονται από την κρίση με προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων ευρώ. Πολλές αντιπροσωπείες της Ένωσης έχουν διοργανώσει ε, ημερίδες ανοιχτών θυρών ε, για να εορτάσουν τη 15 η επέτειο από το ψήφισμα 1325, έρχονται σε επαφή με τοπικές ομάδες γυναικών, το χάρη στη Βοσνία Ρεζεγοβίνη, στο Ιράκ, στο Κωσυφοπεύσα μέσα Οκτωβρίου και η Αφρικανική Ένωση μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση διοργάνωσε ένα σεμινάριο στην Αντίσα για τις γυναίκες με στόχο τη διατύπωση συστάσεων για κοινέ δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης και σε ό,τι αφορά τις ε, δεσμεύσει ε, που μπορούμε να ανανεώσουμε και να υπολογίσουμε, να μετρήσουμε, προβλέπουμε πριν από τα τέλη του έτους να εκπονήσουμε ε, κάποια προγράμματα εκπαίδευση για τα δικαιώματα των παιδιών, των γυναικών για την εκπαίδευση του προσωπικού των αντιπροσωπιών ε, σε θέματα ΚΕΠΑ. Και για το 2013 θέλουμε να αναπτύξουμε τοπικές στρατηγικές ε, για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 σε ό,τι αφορά την αναπτυξή συνεργασία σε τουλάχιστον το 60% των χωρών ε, που είναι σε κατάσταση σύγκρουσης ή έχουν μόλις βγει από μια τέτοια κατάσταση. Έχουμε λοιπόν σταθερή δέσμευση, έχουμε 17 δείκτες οι οποίοι εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2013 2010 και ε, όπου να είναι θα ολοκληρωθεί και η πρώτη έκθεση για τη συνήκη και την ασφάλεια. 26 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε σε μια συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, ε, επί τη ευκαιρία της 10 η επαιτίου από το ψήσμα 1325 και προηγουμένω είχε διοργανώσει τρει εκδηλώσει η Βελγική Προεδρία σε υπουργικό επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων στι Βρυξέλλε, τη Νέα Υόρκη και τη Γενέβη για να ευαισθητοποιήσει και για να διατυπώσει συστάσει. Επομένω η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά συνηγορεί και ζητά να υπάρχει διεθνή παρακολούθηση για την εφαρμογή του ψηφίσματο 1325 ιδίω τονίζοντας όλους αυτούς τους δείκτες ε, που έχει αναπτύξει ο Γενικός Γραμματέας. Καλή λοιπόν τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, σωστή εφαρμογή των ε, δικτών αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας εκ μέρους του Συμβουλίου. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Χωακίν Αλμούνια. Ποιος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τη Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου για τα λόγια της σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια τα στηρίζει πλήρως. Στηρίζει πλήρως τα όσα είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Και θέλω εγώ να προσθέσω τρεις συγκεκριμένες πτυχές. Καταρχάς, θέλω να επισημάνω ότι συμφωνώ πλήρως με αυτό που είπε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου υπάρχει σαφής πρόοδος με πάνω από 20 εθνικά σχέδια δράσης τα οποία υλοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, πρώτος ειδικό εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των γυναικών σε ένοπλε συγκρούσει, ο ορισμός αυτός είναι επίσης ένα σημαντικό γεγονός. Και θέλω επίσης να σας πω το εξή. εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε ένοπλες συγκρούσεις και ιδίως κατά της σεξουαλικής ή ε, βίας που σχετίζεται με το φύλλο, κάτι που καταστρέφει τη ζωή πολλών ατόμων. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να, όπως είπαμε, να εφαρμόσει το ψήφισμα 1325 και τα άλλα ε, ψηφίσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να δίνουμε προσοχή στις ανάγκες των γυναικών, των κοριτσιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις. Επίσης, ε, και σε, μετά από ένοπλες συγκρούσεις καταστάσεις μέσω προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούν του παραδείγματο χάρη παροχή ιατρικών ε, υπηρεσιών ε, για θύματα σεξουαλικής ε, βίας μέσω ομαδικής εργασίας με την κοινωνία των πολιτών για να ευνοήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Και βέβαια συνεργαζόμαστε στενά και με το Ηνωμένα Έθνη για την κατάρτιση των δικτών που η Γενική Γραμματεία έχει αναπτύξει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει και άλλα βήματα. Παραδείγματο χάρη, η αντιπρόεδρος ε, και ύπατη εκπρόσωπος ε, Κάθριν Άστον έχει ορίσει την πρώτη γυναίκα ειδική εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σουντάν, την κυρία Ρόσελιν Μάρσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, για τις παρατηρήσεις σας. Εξ ονόματος τώρα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η κυρία Έντιτ Μπάουερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το 1325 που ευθύθηκε πριν από μια δεκαετία ήταν ένα σημαντικό βήμα που ελήφθη μετά από τις εμπειρίες που είχαμε στον πόλεμο στην πρώην αυτά οι οποίοι υποφέρουν ε, όσον αφορά τον ε, άμαχο πληθυσμό σε κάποιον πόλεμο είναι κυρίως οι γυναίκες. Οι ένοπλες συγκρούσεις συχνά συμπεριλαμβάνουν ε, και το βιασμό γυναικών ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα όσα αναφέρει και η συνθήκη της Γενέβης σχετικά. Επίσης, συνέπειες αυτές συχνά καθιστούν τη ζωή μετά τη σύγκρουση αδύνατη καθώς η σωματική και ψυχολογική ταπείνωση αφήνει τα ίχνη σε μια ολόκληρη ζωή αν υποθέσουμε πρώτα απ' όλα ότι θα καταφέρει να αναρρώσει το θύμα. Οπότε θα πρέπει η πρόληψη της βίας κατά των ε, γυναικών να γίνει μέρος της ε, ευρωπαϊκής εξωτερικής ε, πολιτικής για να μπορέσουμε να προλάβουμε τέτοιες πράξεις. Προφανώς δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον ΟΗΕ εδώ πέρα. Κάτι πρέπει να προκύψει από αυτό, γιατί ακόμα και σήμερα βιάζονται κατά οι γυναίκες και μετά εξωστρακίζονται από τις οικογένειές τους, οπότε θυματοποιούνται για δεύτερη φορά. Μην ξεχνάτε πως στο Κονγκό 830.000 βιάστηκαν σε μία πενταήμερη περίοδο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι συμβαίνει λοιπόν και στην Αφρική και στα στρατόπεδα εκείνα που δεν ζουν με ασφάλεια οι γυναίκες. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στις ειρηνευτικές δυνάμεις γιατί η παρουσία γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντική. Θεωρούμε πως είναι σημαντικό για τις γυναίκες να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαδικασίες. Δεν μπορούν να παίζουν μόνο το ρόλο του θύματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Εξονόμαστος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Μαρία Ελένη Κοπά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμπληρώνονται 10 χρόνια από το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Και είναι μια σημαντική επέτειος, πιο επίκαιρη από ποτέ γιατί οι γυναίκε, όπω και τα παιδιά είναι ακόμα τα μεγαλύτερα θύματα των πολεμικών συγκρούσεων. τα χιλιάδε κρούσματα βιασμού στι εμπόλεμε περιοχέ αποδεικνύουν ότι οι βιασμοί και η σεξουαλική κακομεταχείριση χρησιμοποιούνται συστηματικά ω πολεμικό όπλο για την ταπείνωση και εκμηδένιση του ηθικού του αντιπάλου. σε πολλέ περιπτώσει, οι στρατιώτε, καθοδηγούμενοι από του ανωτέρου του, προχωρούν συστηματικά σε βιασμού, οι οποίοι αν είναι δημόσιοι είναι ακόμα μεγαλύτερο το πλήγμα στον αντίπαλο τα θύματα των πρακτικών αυτών κατά κανόνα γυναίκες στιγματίζονται απορρίπτονται ή ακόμα και δολοφονούνται από την ίδια την κοινότητά τους στην προσπάθεια να αποκατασταθεί η τιμή. πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε αυτή τη μάχη να σταματήσει αυτό το έσχος για την ανθρωπότητα αυτά τα εγκλήματα πολέμου. πρέπει παράλληλα να αυξήσουμε τους ελέγχους παντού και μεταξύ των γιανόκρανων, γιατί και οι δικές τους ευθύνες άμεσες ή έμεσες είναι μεγάλες. απαιτείται η έμεσε ειναι μεγαλες αυστηρών κυρώσεων σε όσους εμπλέκονται σε τέτοιες πράξεις χρειάζεται εκπαίδευση έλεγχος και αυστηρότητα και ξεκάθαρο μήνυμα. τελικά πρέπει να δείξουμε ως διεθνή κοινότητα ότι εννοούμε αυτά που λέμε. οι γυναίκες όπως λέει το ψήφισμα 1325 μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα στην προώθηση της ειρήνης και ασφάλειας. στόχος όλων μας πρέπει να είναι να ενδυναμωθούν οι γυναίκες με δυνατότητα προσφυγή σε διεθνή δικαστήρια με προγράμματα για την οικονομική κοινωνική και ψυχική επανένταξή του η χειραφέτησή τους και η προστασία τους είναι ο αναγκαίος όρος για να μπει ένα τέλος στη χρήση της σεξουαλικής βίας ως όργανο πολέμου. ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Η κυρία ο Λάι από τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες. Δεν είναι παρούσα. Από ό,τι βλέπω, δηλαδή είναι απούσα. Από τους Πρασίνους, η κυρία Μπάρμπαρα Λόχμπιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώντας ε, δικαιοσύνη για τα φύλλα στε περιοχές πολέμου πριν από 10 χρόνια <laughs> έγιναν για πρώτη φορά αυτά τα ζητήματα θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ένα ορόσημο για να οδηγηθούμε σε δεσμευτικές ε, διατάξεις στη συμπερίληψη αυτών των θεμάτων στην ε, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Και το 2005 ο Κόφι Ανάν ζήτησε κατεπηγόντως εθνικά σχέδια δράση για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325. Ακούσαμε ήδη πως αυτό το έκαναν μέχρι τώρα μόνο 20 χώρες, μεταξύ των οποίων ευρωπαϊκές όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Σουηδία, αλλά και αφρικανικές χώρες όπως η Λιβερία και η ακτή του Ελεφαντοστού. Και θεωρώ πως απαιτείται από όλα τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν τέτοια σχέδια δράσης, χώρες όπως και η δικιά μου η Γερμανία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει υποβάλει ένα τέτοιο σχέδιο δράσης. Η δε προοπτική του φίλου έχει κερδίσει σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχει νέος ε, ειδικό αποσταλμένος του ΟΗΕ για τις ε, γυναίκες και για την ισότητα, αλλά αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι ακόμα στην αρχή. Το θέμα είναι η υποστήριξη των θυμάτων εδώ πέρα. Έχουμε προγράμματα βοήθειας που πρέπει να εντετικοποιηθούν, αλλά το θέμα είναι και η υποστήριξη και της ποινική δίωξη των δραστών. Και βεβαίως αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρξει και επιτόπου μεταρρυθμίση της ε, δικαιοσύνης. Θετικό είναι αυτό το οποίο είπε ο πρόσωπος της της ε, ε, Άστον πως θα πρέπει να υπάρξει με χρηματοδότηση 200 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί το ψήφισμα αυτό και θα ήθελα να υπενθυμίσω πόσο αναγκαίο είναι να ενισχύσουμε τις τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα λεφτά στοχευμένα. Ευχαριστώ κυρία Εύα Μπριτ από την Ενωμένη ΕΕ. Ευρωπαϊκή Αριστερά. Σας ευχαριστώ. Οι γυναίκες συνήθως είναι θύματα στις, ε, στις ε, καταστάσεις ε, της εμπόλεμες. Χρησιμοποιείται όπλο, ως όπλο η βία κατά των γυναικών και των παιδιών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι γυναίκες λοιπόν είναι θύματα. Να θυμίσουμε τα όσα είπε ο ειδικό απεσταλμένος του ΟΗΕ. Μα οι γυναίκες δεν είναι μόνο θύματα, είναι και σημαντικοί παράγοντες όσον αφορά την διατήρηση της ειρήνης και τη σχετική εργασία, καθώς και στην δουλειά, στην εργασία της πρόληψης των συγκρούσεων. Είναι πολύ σημαντικές για την οικοδόμηση της δημοκρατίας μετά από τους πολέμους και τις συγκρούσεις. Πολύ σημαντικές για την ανοικοδόμηση των χωρών. Δέκα χρόνια μετά την έγκριση του ψηφίσματος του ΟΗΕ 1325, ακόμα σήμερα σήμερα οι γυναίκες ε, μόνο θεωρούνται θύματα της βίας, αλλά δεν ε, γίνεται αντιληπτή η σημασία της όσον αφορά την ανοικοδόμηση μετά από τον πόλεμο, μετά από τη σύγκρουση και την ε, διατήρηση της ειρήνης. Είναι αλήθεια πως οι γυναίκες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν, αλλά τελικά οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους άνδρες. Οι ικανότητες των γυναικών για την στην, στο στο, στο πλαίσιο μια, της ερευνητικής διαδικασίας θα πρέπει να αξιολογηθεί, να αξιοποιηθεί. Θα πρέπει αυτό να το σκεφτούμε, σκεφτόμαστε πάντα. Ευχαριστώ. Της ε, ομάδας Ευρώπη Ελευθερίας Δημοκρατίας, ο κύριος Πάσκα, για 1,5 λεπτό το λόγο. Rezolúcia číslo 1325 Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov o ženách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 συχνά οι πολιτισμένες χώρες ε, προσπαθούν να επιβάλλουν τα όσα αναφέρονται στο ψήφισμα 1325 και να δημιουργηθεί ένα δεύτερο πλαίσιο για την ε, εφαρμογή τους. προβλήματα τα οποία πρέπει να ληφθούν ε, σοβαρά υπόψη ε, για το σεβασμό των γυναικών υπάρχουν και στην Κεντρική Αφρική και σε κάποιες ασιατικές ε, χώρες. Ξέρετε πως τα στρατιωτικά καθιστώτα βασίζονται σε τελείως διαφορετικές αξίες από αυτές που αναγνωρίζει η δική μας κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν πως θα πρέπει πρώτα απ' όλα να επικεντρωθούμε σε αυτόν τον τομέα Πρέπει να λάβουμε μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη πίεση σε καθεστώτα τα οποία παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων τους. Τώρα για το από την ομάδα των μη εγγεγραμμένων η κυρία Μορβάουη για 1,5 λεπτό θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω πως όλοι θα μπορούσαν να δώσουν μια εύκολη απάντηση στο ερώτημα του ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες λαμβάνουν τις οικονομικές ή τις πολιτικές αποφάσεις. Όμως, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ε, αυτή είναι και που ε, θα πρέπει να σκεφτούμε ποιε είναι οι ομάδε που φέρουν τι συνέπειε αυτών των αποφάσεων, ειδικά όταν μιλάμε για θέματα όπω τα σημερινά, όταν μιλάμε για την οικονομία. Οι γυναίκε είναι αυτές που πρέπει να φέρουν το φαγητό στο τραπέζι των οικογενειών του. Αυτές είναι που υποφέρουν από τη φτώχεια μαζί με τα παιδιά του, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε. Και αν δούμε τις συνέπειες ε, των, ε, του ψηφίσματος ε, του ΟΗΕ, οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν περισσότερο χώρο, περισσότερο ρόλο να παίξουν ε, μεγαλύτερο ρόλο να παίξουν συγγνώμη, στις, ε, στη λήψη των αποφάσεων, γιατί αυτές είναι που επηρεάζονται περισσότερο. Επηρεάζονται και από τις εμπόλεμες σειράξεις, ε, από τις ένοπλες σειράξεις. Κοιτάξτε στη Γάζα, για παράδειγμα, τι γίνεται. Οι γυναίκες είναι αυτές που φροντίζουν τους τραυματισμένους μετά από τις βίες επιθέσεις του Ισραήλ. Εκείνες που φροντίζουν τα παιδιά που πρέπει να ζήσουν ανάπηρα την υπόλοιπη ζωή τους. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, επαναλαμβάνω, οι γυναίκες είναι που ασχολούνται ε, και βλέπουμε ότι οι βόμβες καταστρέφουν σχολεία, δρόμους. Πρέπει όλα αυτά να τα σκεφτούμε όταν μιλάμε για τις ε, γυναίκες ε, θύματα ως αποτέλεσμα των ενόπλων σειράξεων. Των άλλων εγγεγραμμένων μιλητών. Ε, τώρα θα πάρει το λόγο ο κύριος Ζιβάν για δύο λεπτά παρακαλώ. Monsieur Juvin. Madame la Présidente, Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, στις ε, εμπόλεμες περιοχές η βία κατά των γυναικών εγγράφεται στο πλαίσιο μιας ηθελημένης τακτικής. Ε, ο βιασμός είναι μαζική πρακτική, συστηματική και σχεδιασμένη, προγραμματισμένη πρακτική, είναι όργανο πολέμου. Και βέβαια θα πρέπει να καταδικάσουμε αυτές τις πράξεις βίας. Πέραν της καταδίκης όμως, οι δηλώσεις, τα λόγια δεν επαρκούν. Αλλιώς πρέπει να προχωρήσουμε σε, μάλλον διαφορετικά σε συγκεκριμένε πίστε δράσεις. Και θα έλεγα προ τρει κατευθύνσεις, κύριε Πρόεδρε. Πρώτη κατεύθυνση, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι σε κάθε ένοπλη σύγκρουση, όπου και αν συμβαίνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθεί τις τοπικές γυναικέ οργανώσεις. Ο σεβασμός των βασικών πρακτικών ελευθερίας και δικαιοσύνης θα ενισχυθούν εάν βασίζονται, αν στηρίζονται στις γυναίκες παντού όπου δίνουμε στον κόσμο δικαιώματα στις γυναίκες, ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ο σεβασμός ε, της αδελφότητας, της αδελφοσύνης ε, και των αρχών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης προοδεύουν. Δεύτερη πίστα, δεύτερη κατεύθυνση, όταν εμείς Ευρωπαίοι συμμετέχουμε στην ενίσχυση προς υποδόμηση χώρες, νομίζω ότι θα πρέπει να απαιτήσουμε από τους ηθήνοντες, από την τοπική αυτοδίκηση επιτόπου, να εφαρμόσουν ποσοστώσεις, δηλαδή συμμετοχή γυναικών στα κρατικά εξώματα. Παραδείγματος χάρη στην Παλαιστινιακή Αρχή που έχουμε 100% σχεδόν χρηματοδότηση εκ μέρους μας θα πρέπει νομίζω ότι σε θέσει ευθύνη, πολιτική ευθύνη, να προωθήσουμε τι ποσοστώσει ε, γυναικών. Μόνο ωφελημένη θα είναι η περιοχή από αυτό. Τρίτη ε, σκέψη, όπου παρεμβαίνουμε ε, είτε με στρατιωτικό, είτε με μη στρατιωτικό τρόπο, είτε μέσω αστυνομία. Νομίζω ότι θα πρέπει να δεσμευτούμε ένα σημαντικό μέρο, προσαρμοσμένο βέβαια και στι συνθήκε, να το εκχωρήσουμε στι γυναίκε, δηλαδή και στα στρατεύματα ε, και στι επιχειρησιακέ μονάδε, να υπάρχει επαρκή αριθμό γυναικών. Έτσι θα είναι πιο αποτελεσματικέ οι μονάδε αυτέ και θα είναι αποδεκτέ και από τον τοπικό πληθυσμό, όπω δείχνουν και πολλέ μαρτυρίε. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριο Ταραμπέλα για δύο λεπτά επίση. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και δέκα χρόνια ενέκρινε για πρώτη φορά το Συμβούλιο Ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών ένα ψήφισμα που τονίζει την ειδική κατάσταση των γυναικών σε εμπόλεμε περιοχέ και για την επίλυση των συγκρούσεων. Μετά από 10 χρόνια εξακολουθούν να βιάζονται οι γυναίκε σε εμπόλεμε περιοχέ όπω το Κονγκό, για παράδειγμα. Εγώ έχω καταδικάσει την ατιμορρησία τη οποία χαίρουν οι δράστε εδώ και χρόνια και πέραν αυτού αυτέ οι βαρβαρότητε λαμβάνουν χώρα ε, ενώ υπάρχουν επιτόπου και στρατεύματα του ΟΗΕ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη πολιτική, κατάλληλη χρηματοδότηση, θα πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό ε, των ευρωπαϊκών αλλά και των διεθνών οργανισμών, να ευαισθητοποιηθούν οι πληθυσμοί. Η πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά για να σας παρακολουθούν οι Ευχαριστώ βεβαίως κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι η συνειδητοποίηση της ευθύνη ε, διάστασης του φύλου θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς και θα πρέπει να σταματήσει ατιμορρησία ε, για τη βία κατά των γυναικών και θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες δομές. Θα πρέπει επίσης να αυξηθούν οι χρηματοοικονομικοί πόροι ε, των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για τις εργασίες σε θέματα φύλου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως για την εκτέλεση των μηχανισμών και την αξιολόγηση της προόδου της Ευρωπαϊκής είπε και ο επιτευχθεί πρόοδη, ιδίω στον τομέα τη ανταλλαγή καλών πρακτικών, μέσω τη συμμετοχή σε μια task force. Επίση, πάνω από 10 ε, χώρε έχουν πλέον εθνικά σχέδια δράση και ελπίζω και οι άλλε 17 να κάνουν γρήγορα το ίδιο. Εγώ πραγματικά ε, έχω το, να τι ελπίδε μου στη μελλοντική υπηρεσία εξωτερική δράση. Ελπίζω να βοηθήσει στην ισότιμη παρουσία δρόμων και γυναικών, ιδίω επιτόπου ε, και βέβαια στο ε, ψήφισμα για την επίλυση των συγκρούσεων θα πρέπει να μιλήσουμε για ε, την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των, ε, του προσωπικού των εργανώσεων και του τοπικού πληθυσμού. Κύριε Φιγκερέιτλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε τις επιπτώσεις των πολέμων και των συγκρούσεων στα παιδιά και στις γυναίκες σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή όπως αυτή που διανύουμε, όπου μένονται οι πόλεμοι στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, τροφοδοτούνται σοβαρές συγκρούσεις στα κατεχόμενα εδάφη της Παλαιστίνης, στην Δυτική Σαχάρα ή από το Μαρόκο. Πολλαπλασιάζονται οι ανισότητες και αυξάνεται η φτώχεια μέσω των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Δημιουργούνται νέα προβλήματα όπως διαπιστώσαμε στη Λισαβόνα αυτή την εβδομάδα με το ενδιάσκεψη κορυφή του ΝΑΤΟ και την υιοθέτηση της νέας ε, στρατηγική του, του νέου στρατηγικού του δόγματο. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ τη εκστρατεία, ε, ε, ειρήνη ναι και εκεί διαδήλωσαν ε, χιλιάδες άνθρωποι υπέρ της ε, ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ασφάλειας και φώναξαν ε, κατά του ψηφίσματος του ΝΑΤΟ υπέρ της του πυρηνικού αφοπλισμού. Αύριο η γενική απεργία που θα γίνει στην απεργία θα κινητοποιήσει και εκ νέου γυναίκες και άνδρες που πολεμούν τις αντικοινωνικές πολιτικές και οι οποίες ιδιαίτερα ασκούν διακρίσεις κατά των γυναικών αλλά και κατά κατά των, και υπέρ των πολιτικών που σέβονται αυτούς που εργάζονται και που προωθούν την κοινωνική πρόοδο, που είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ βεβαίως ε, Χαιρετίζω το ψήφισμα 1325. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την ειρήνη και την ειρηνευτική πολιτική. Ήταν η πρώτη φορά κατά την οποία ο ΙΕ αναγνώρισε την σημασία της ε, πρόληψης ε, των συγκρούσεων και των συνεπειών που έχουν στις γυναίκες και θα πρέπει να επιδειχθούν οι στόχοι του. Παρ' όλα αυτά, μετά από δέκα χρόνια η βία εις βάρος ε, των γυναικών αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά των ε, συγκρούσεων όλο και πιο συχνά οδηγούμαστε σε συστηματική βία κατά των γυναικών κατά τη διάρκεια και των συγκρούσεων και μετά από αυτές. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω συγκεκριμένα νούμερα. Ξέρετε τι έχει συμβεί στον Ταρφούρ, στο Κονγκό, στη Ρουάντα, στη Λιβερία, Σιέρα ή στη Βοσνία. Εγώ προσωπικά έχω συναντήσει πολλές γυναίκες που ήταν θύματα βιασμού στην ε, πρώην Γιουγκοσλαβία και οι αναμνήσεις τους είναι τρομακτικές. Βιάστηκαν, βασανίστηκαν, ε, αποκλείστηκαν από την κοινωνία. Το τέλος λοιπόν μια σύγκρουσης δεν σημαίνει πως ε, έχουν τελειώσει και τα βάσανα μιας γυναίκας. Οπότε η προστασία των γυναικών και η συμμετοχή τους στην οικοδόμηση της ειρήνης και της ασφάλειας και αυτά περιέχονται στο ψήφισμα 1325. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ πως υπάρχει μια πραγματική δυνατότητα να τελειώσουν όλα αυτά. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για να δημιουργηθούν οι σωστές συνθήκες για όλα αυτά. Εκπληρώντας αυτές, ε, αυτή την αποστολή θεωρώ πως ε, θα μπορέσει η κυρία Στον να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και η εξωτερική υπηρεσία της άλλωστε. Τώρα το λόγο θα πάρει για ένα λεπτό η κυρία Λέσινγκ. Ευχαριστώ. Οι γυναίκες και τα παιδιά εξακολουθούν σε δυσανάλογο βαθμό να υποφέρουν από τον πόλεμο. Δεν μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν για να νομοποιηθούν στρατιωτικές παρεμβάσεις. Το παράδειγμα του Κονγκό καταδεικνύει πως ε, οι στρατιωτικές παρεμβάσεις δεν συνεισφέρουν σε διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Δυστυχώ διαπιστώνουμε ότι συμβαίνει το αντίθετο στο Αφγανιστάν. Η θέση των γυναικών μέσω του πολέμου έγινε χειρότερη. Η υπόσχεση του ψηφίσματος 1325 μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της αποφυγής των συγκρούσεων και των πολέμων και της χρήσης πολιτικών μέσων. Γι' αυτό δεν νομίζω πως είναι σωστό να καταλήξουμε να λέμε από το ψήφισμα αυτό πως πρέπει να αυξηθεί η παρουσία γυναικών στα πεδία των μαχών θα πρέπει να υπάρξει νομίζω μια καλύτερη εκπαίδευση και των καθεστώτων και των ενόπλων των καθεστώτων τα οποία είτε στέλνουν αμάχους και παιδιά στο πεδίο της μάχης είτε χρησιμοποιούν τις γυναίκες κατά αυτόν τον τρόπο. Η δικασία έχουν ζητήσει να παρέμβουν τέσσερις συνάδελφοι. κυρία Στρέλα. Κύριε Κύριε Πρόεδρε, ήδη αναφέρθηκαν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ε, τα σχέδια ε, στήριξης και υπογραμμίστηκαν ε, τα στοιχεία. Όμως η αλήθεια είναι πως οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν τα μεγαλύτερα θύματα των ενόπλων σειράξεων. Είναι θύματα, αλλά δεν λαμβάνουν αποφάσεις. Οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία της πρόληψης και της επίλυσης των συγκρούσεων. Αν υπήρχαν περισσότερες γυναίκες στις υψηλές θέσεις ε, τις πολιτικές αλλά και στις ε, θέσεις λήψης οικονομικών αποφάσεων θα υπήρχε περισσότερη ειρήνη και ασφάλεια στον κόσμο και όλοι μας ε, θα χαίραμε μεγαλύτερη εξέλιξης, ανάπτυξης και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται περισσότερες γυναίκες στη λήψη των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα όπως ήδη υπόθηκε επανειλημμένως, οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν, θα πρέπει να είναι φορείς, ε, παράγοντες όλη αυτή τη διαδικασία που δεν θα πρέπει απλώς να διεξάγεται από τους άνδρες. Σας ευχαριστώ. πολύ κυρία Στρέλα. Η κυρία Παρβάνοβα έχει το λόγο τώρα. Κυρία Πρόεδρε, όταν μιλάμε για γυναίκες σε εμπόλεμες ε, περιοχές θα πρέπει να δούμε ότι έχουν γίνει ήδη προσπάθειες όπως από τη Μάργκοτ Μάσον, πρώην επίτροπο που είναι ειδική απεσταλμένη για τη σεξουαλική βία στις ε, συγκρούσεις ε, του ΟΗΕ. Χρειάζεται περισσότερη δράση, μεγαλύτερη συνειδητοποίηση καθώς και συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες στον τομέα αυτό. Να τονίσω πως συνεργασία ανάμεσα στους βουλευτές στις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των ΗΠΑ καθώς και η συνεργασία στην κοινωνία των πολιτών είναι βασικές για την προάσπιση αυτών των στόχων σε διεθνή πλαίσια καθώς και για την ανάπτυξη των στόχων της χιλιετίας. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δεσμευθούμε από κοινού και να προωθήσουμε το ζήτημα εξασφαλίζοντας καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στην προσπάθεια ε, στις εμπόλεμες περιοχές αλλά και στις ε, ε, καταστάσεις μετά από πολέμους καθώς οι γυναίκες μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και στην ε, εξασφάλιση της ειρήνης. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κρίσιμο ρόλο να παίξει στην πρόθεση αυτών των στόχων ώστε να επιτευχθεί μια ισότιμη και διαρκής λύση. Αυτή είναι η κύρια δική μας ευθύνη και σημαντικός πολιτικός ρόλος ε, μας βαραίνει όσον αφορά την υπεράσπιση των γυναικών και τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία uh, um, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να εκφράσω τη στήριξή μου για το ψήφισμα 1325 ε, και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στη Βόρεια Ιρλανδία όπου έχουμε πολύ δραστήριο γυναικείο τομέα. Έναν τομέα που έχει ενισχυθεί και έχει εμπεδοθεί στην χώρα. Εγώ αντιπροσωπεύω το, αντιπροσωπεύω το δυτικό Μπέλφαστ στην ε, Βουλή της Βόρειας Ιρλανδίας. Είναι περιοχές που έχουν ε, υποφέρει από 30 χρόνια βίας. Είχαμε ε, τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο IRA αλλά και ενδοκινοτικές συγκρούσεις και ολόκληρο εκείνη την περίοδο οι ομάδες όπως το η Women Center είχαν μια πραγματική ισχύ και ενίσχυσαν τους δεσμούς με με άλλες ε, γυναικείες ε, κοινότητες. Ε, είναι απλές γυναίκες που απέδειξαν ότι είχαν ηγετικές ικανότητες, απέδειξαν ότι μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν σε βίαιη και ε, κατάσταση. Σήμερα λοιπόν έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχα δίκτυα και προχωρούν, προοδεύουν όσον αφορά τη βελτίωση των κοινοτικών σχέσεων στην Βόρεια Ιρλανδία, αλλά δημιουργούν και ευκαιρίες στην αγορά εργασίας μέσω της παιδείας και της κατάρτισης. Αυτός είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε, συνάδελφοι. Νικολάου θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Uh, Ευχαριστώ. πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ και ελπίζω η σημερινή συζήτηση πως δεν θα είναι μόνο μια, ένας εορτασμός της δεκαετούς επαιτίου του 1325 αλλά και ένα κάλεσμα για να λάβουμε δράση καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι αυτή η οποία ήταν πριν από μια δεκαετία. Δεν αρκούν οι δηλώσεις ε, καλής θέλησης βεβαίως πραγματικότητα, ναι, αλλά πρέπει να δράσουμε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ε, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στις ε, επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και μετά τις συγκρούσεις. Υπάρχει λοιπόν ε, και ρήτρα στη συνθήκη της Γενέβης που μιλάει για ποινικοποίηση της βίαιης συμπεριφοράς στις συγκρούσεις. Κάτι το οποίο νομίζω θα ήταν προσθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει να το επιτύχει. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε όλες μας τις δράσεις με τα ανάλογα κονδύλια και να έχουμε μια ενιαία στάση και στην αναπτυξιακή μας πολιτική. Έχετε το λόγο κύριε Ζαμπόσκα. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ξέρετε πως ε, σήμερα έχουμε Γιορτάζουμε την 15 η επέτειο του ψηφίσματο 1325 του Συμβουλίου Ασφαλεία ε, του ΟΗΕ σχετικά με τι γυναίκε, την ειρήνη και την ασφάλεια. Έχω όμω κάποιε ανησυχίε για το εάν πραγματικά ελέγχουμε σοβαρά την εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος. Η κατάσταση βελτιώνεται πάρα πολύ αργά. Είναι υποχρέωσή μα να βοηθήσουμε τις ε, γυναίκες να ενσωματωθούν στην ε, κοινωνία ανεξαρτήτως από την ε, προέλευσή τους. Αυτό ξεκινάει ήδη από την οικογένεια. Η οικογένεια είναι υπεύθυνη για την ανατροφή των παιδιών και θα πρέπει βεβαίως να μπορούν να ζουν οι γυναίκες χωρίς ταπείνωση και οπωσδήποτε πολύ περισσότερο στον ε, πόλεμο. Επιπλέον, εάν δεν μπορεί κάποιος να αισθάνεται ασφαλή στην οικογένεια και στην πατρίδα του, δεν μπορούμε να μιλάμε για ειρήνη. Και το λόγο θα πάρει ο Υπουργός ο κύριος Σατέλ, εξ ονόματος της είπα της εκπροσώπου της κυρίας Άστον. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Φυσικά και συμφωνώ με πάρα πολλά από όσα είπαν ε, οι ευρωβουλευτές. Πώς μπορεί κανείς να μην συμφωνεί με αυτό που ο κύριος Ζιβά, ο κύριος Ταραμπελά για τον τρόπο με τον οποίο η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης πρέπει να αποτελέσει μείζωνα ευκαιρία για ενδυνάμωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Στη διαδικασία της ε, υλοποίησης της υπηρεσίας αυτής ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μόνιμη πρόκληση καλύτερης γυναικείας εκπροσώπησης σε όλα τα επίπεδα και ε, στο προσωπικό και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Η Λέδη Άστον πραγματικά ε, πηγαίνει προς την κατεύθυνση αυτή με σαφή μέτρα. Παραδείγματο χάρη έχει ορίσει την πρώτη εκπρόσωπο, την κυρία Ρόζαλιν Μάρστιν ως ειδική εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σουδάν. Το Σεπτέμβριο 29 γυναίκες έχουν καταλάβει θέσεις στη διοίκηση και τα γυναίκες είναι επικεφαλής διοικήσεων. Ε, Αυξημένο αριθμό λοιπόν γυναικών που είναι παρόντες στα υψηλά αυτά αξιώματα και επίση ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τι δυνατότητε τη και τι ικανότητέ τη για την ε, για τομέα των γυναικών της ειρήνης και της ασφάλειας. Και βέβαια θα πρέπει επίσης να ευαισθητοποιήσουμε και άλλες οργανώσεις, άλλους οργανισμούς, άλλες χώρες και αυτό βέβαια ε, πηγαίνει χέρι-χέρι με ειδικέ εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Πολύ το σχολιάσατε αυτό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ε, Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, για την υλοποίηση του ψηφίσματος σε χώρες όπως το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, Γεωργία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και η κοιλάδα το Φεργκάνα, Ουσμπεκιστάν, Κυργιστάν και τα Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί θα θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη επευθυνότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συμβούλιο Ασφαλεία θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα εργασία που θα εξετάσει ε, την πρόοδο που έχει επιτελεστεί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ψηφίσματο 1325 και επίση θα πρέπει να διατυπώσει συστάσει στο Συμβούλιο για να μετοπιστούν τα κενά, οι προκλήσει και να επιταχυνθεί η υλοποίηση του ψηφίσματο. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλεία ε, να πολλαπλασιάσει τι προσπάθειέ του στον τομέα τη καταπολέμηση λέμε της ατιμορρησίας. Ε, ε, στοχευμένα και σταδιακά ε, μέτρα και κυρώσεις που θα πρέπει να επιβληθούν σε όσους διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων γυναικών. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια και των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, έλαβα έξι προτάσεις ε, ψηφίσματος από αντίστοιχες πολιτικές ομάδες για το θέμα αυτό της συζήτησης. Έληξα όμως εδώ η συζήτησή μας και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, 5η στις 12 το μεσημέρι. Τώρα ερχόμαστε.